ψηφοφορία θα λάβει χώρα στη συνέχεια. Ακολουθεί η ψηφοφορία για έξι ψηφίσματα για την Βενεζουέλα. Δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες. Ε, υπάρχει κοινό ψήφισμα ε, τριών πολιτικών ομάδων. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι είναι άλλοι τρεις συνάδελφοι. Ε, ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Το ψήφισμα εγκρίνεται με 41 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 3 αποχές. Ε, βάσει της ημερήσιας διάταξης ακολουθεί η ψηφοφορία για έξι ψηφίσματα για τη Ματαγασκάρ. με ένα κοινό ψήφισμα έξι πολιτικών ομάδων. Δεν έχουμε προτροπολογίε. Θα ψηφίσουμε με απλή ψηφοφορία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Με λίγες αποχές εγκρίνεται ομόφωνα ε, το ψήφισμα. Τώρα, έξι ψηφίσματα για τη Βυρμανία. Υπάρχει ένα ε, κοινό ψήφισμα έξι πολιτικών ομάδων και δύο συναδέλφων. Τροπολογία υπαρθμών 1 για την παράγραφο 14. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα θα έχουμε συνολιστική ψηφοφορία για το ε, ούτως τροποποιηθέν ε, σχέδιο ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται ομόφωνα και χωρίς αποχές. Τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης θα υποβληθούν στην προσεχή συνεδρίαση προς έγκριση. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, ε, λύεται η συνεδρίαση. Διακόπτονται οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η συνεδρίαση Ολομέλειας, λύεται η συνεδρίαση. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.